Υπάρχει σοβαρός κινδύνος, κυρία Νταλάρη, να ε, θανατωθεί. Και εξ ονόματος όλων θα επαναλάβω την εκκλησία μου προς τις αρχές της Τεχεράνης για να μην εκτελέσουν την ποινή. Εξ ονόματος του Κοινοβουλίου ε, καταδικάζουμε την θανατική ποινή σε οποιαδήποτε περίσταση γιατί αντίκειται στις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Κιέγγε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να θυμίσω την φρικτή κατάσταση της ε, Περιοχή μου, τη Εμίλια Ρωμάνια, ε, με τι πλημμύρε των ποταμών λόγω των αντίξεων καιρικών συνθήκων. Η κακοκαιρία που έχει πλήξει όλη την Ευρώπη και επειδή τώρα το Κοινοβούλιο ε, στέκεται κοντά στις διάφορες πληγήσει περιοχέ να σταθεί κοντά και στου πληγέντε πληθυσμού εξαιτία των αντίξεων καιρικών συνθήκων και να το εκφράσει αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ενώνω τη φωνή μου στη δική σα, όχι μόνο ω Ιταλό, αλλά και ω πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Ε, είναι δίκαιη η ανησυχία σα, και είμαστε στο πλευρό των ευρωπαϊκών πληθυσμών που επλήγησαν τι τελευταίε εβδομάδε από τι αντίξωε συνθήκε. Την περασμένη εβδομάδα, ε, να θυμίσω τον ε, ρόλο ε, του ε, πρόεδρου της Ρουμανίας που του πρώην βασιλιά της Ρουμανίας, ο οποίος ε, είχε σημαντικό ρόλο στο να προσεγγίσει η χώρα αυτή το σωστό στρατόπεδο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να εκφράσω την, ε, και να τον τιμήσουμε για τον σημαντικό ρόλο που είχε. Ε, κυρία Φορέντσα, να ενημερώσω του συναδέλφου ότι την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην Άγκυρα για να παραστώ στην δίκη δύο πρόεδρων του ΑΚΤΠ. Και να πω ότι δεν μπορέσαμε να έχουν πρόσβαση στην αίθουσα του δικαστηρίου. Μας εμπόδισε η τουρκική αστυνομία. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε τέτοιε καταστάσει ενώ συζητάμε ταυτόχρονα τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Ευχαριστούμε κυρία Φορέντσα για την ε, πληροφορία. Ε, προασπιζόμαστε την ελευθερία και την ε, δίκαιη εκδίκαση υποθέσεων σε όλες τις χώρες και στην Τουρκία.